Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και να καλωσορίσω θερμότατα τον Επίτροπο Έτιγκερ που μας κάνει την τιμή να παρουσιάσει πρώτα στην Επιτροπή μας την ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό του 2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε ε, κύριε Επίτροπε που προτιμήσατε να έρθετε πρώτα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν να κάνετε την ανακοίνωση στον τύπο. Μετά, τη, μετά την απόφαση της, των συντονιστών της 10 η Μαΐου, η σημερινή ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο ε, θα γίνει όσο πιο δυναμικά γίνεται κατ' εφαρμογή του συστήματος ping-pong στοιχομηθεί, δηλαδή. Γιογιό και πινκ πονγκ είναι ορολογία που χρησιμοποιούμε τακτικά στην Επιτροπή προπολογισμών. Οπότε δεν ε, θα ομαδοποιούμε τις ερωτήσεις ε, για να απαντά μαζικά ο Επίτροπος. Αλλά μετά από κάθε ερώτηση θα δίνει αμέσω την απάντηση ο Επίτροπος. Ε, οι ευρωβουλευτέ που υποβάλλουν τις ερωτήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν και συμπληρωματικές επερωτήσεις με σεβασμό όμως ε, στο χρόνο αγόρευσης που δικαιούται ο καθένας. Και μετά την απάντηση, τελική απάντηση του Επιτρόπου δεν θα υπάρχει δυνατότητα ε, να επανέλθει κανείς. Οπότε σας θέρμο παρακαλώ να είστε όσο πιο συνοπτικοί και λακωνικοί γίνεται στην υποβολή των ερωτήσεων, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο ο Επίτροπος για τις απαντήσεις και να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε και επερώτηση μετά την πρώτη απάντηση. Οι διαπραγματεύσεις για τον ετήσιο αυτό προϋπολογισμό θα γίνουν παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε, σε αυτή την έντονη και κατά πάσα πιθανότητα και δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων, είναι σημαντικό να κρατήσουμε ένα ε, σημαντικό σημείο ε, στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή στην ε, απέτηση της εμπιστευτικότητας. Και μάλιστα δύο στοιχεία διέσαν αυτή την ε, εμπιστοσύνη. Καταρχήν η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το μηχανισμό για, τη, για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Το θέμα του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ίσως το αναφέρετε κι εσείς. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων πέρυσι στη συνδιαλλαγή είχαμε ενίσχυση κατά 116 εκατομμύρια ευρώ το προϋπολογισμό το 2018 με βάση μια συμβαστική πρόταση που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις αρχές του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε μια πρόταση που μιλάει για το ίδιο πόσο για το, μέχρι το 2020. Βέβαια είναι ε, ενδεικτική αυτή η πρόταση, δεν είναι δεσμευτική, αλλά ένας ε, έμπειρος πολιτικός σαν και εσάς γνωρίζει ότι αποκλείεται να ευοδοθεί ε, μετά τις διαπραγματεύσεις ε, αυτή η πρόταση δεδομένη της πολιτικής πραγματικότητας. Επιμένω λοιπόν στην ανάγκη της αμοιβέ εμπιστοσύνη. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό για τους πρόσφυγες, ε, το μηχανισμό δηλαδή για την υποδοχή των ασύρων προσφύγων στην Τουρκία, θα μας παρουσιάσετε σήμερα το διορθωτικό προπολογισμό για το μηχανισμό αυτό συμπληρώνοντας τις προτάσεις του 2019. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστηματικά ε, επισήμανε ότι δεν έχει εκτιμήσει ιδιαιτέρως τη θέσπιση αυτού του μηχανισμού και ότι η απόφαση για τη χρηματοδότηση αυτού του μηχανισμού ελήφθη κατά τη γνώμη μας ερήμην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε την αίσθηση ότι πρώτα τα συμφωνείτε με το Συμβούλιο και μετά έρχεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πρόταση του διορθωτικού προϋπολογισμού που ε, οφείλει να εγκρίνει μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θα ήθελα να μας παρουσιάσετε αυτά που κρίνεται σκόπιμα και μετά ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λαμβάνουν θέση. Οπότε υπευλήθη το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού βάσει την αρχική πρόταση με το μοντέλο ότι για 3 δισεκατομμύρια ε, για το μηχανισμό υποδοχής προσφύγων, ε, σύρων προσφύγων στην Τουρκία είχαμε 1 δισεκατομμύριο από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και 2 δισεκατομμύρια από τα συνεισφορά των κρατών μελών μερικές φορές μας κατηγορούν ως εθεροβάμονες οι ουτοπιστές και μπορεί με να έχουμε τα ελαττώματά μας, αλλά εκπροσωπούμε την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε όργανο που εκλέγεται με άμεση και καθολική ε, ψηφοφορία και εκπροσωπούμε επίσης την πολυμορφία, την πολυφωνία και τη διαφορετικότητα. Οπότε και για τον προπολογισμό του 2019 και για το τρίτο διορθωτικό προπολογισμό του 2018 αλλά και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο καλό θα ήταν να αφουγκράζεστε και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι αυτή η εμπιστοσύνη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη θα πριτανεύσει σε όλες τις σχέσεις μας και ε, ελπίζουμε αυτό να συμβεί. Και μάλιστα το σχέδιο που θα μας υπο υποβάλλεται σήμερα είναι το τελευταίο τη τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία και είναι και το τελευταίο παρουσία των Βρετανών συναδέλφων. Του των λεχθέντων, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σα δώσω το λόγο και να επισημάνω ότι είστε διαθέσιμο μέχρι τη μία παρατέταρτο, οπότε θα σας θέρμα παρακαλούσα να μην υπερβείτε το δεκάλεπτο ή το πολύ το τέταρτο στην αρχική σα παρουσίαση. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στο γενικό μας εισηγητή τον κύριο Βιώτη για 7 λεπτά. Έχει δεσμευτεί ότι θα τηρήσει το 7 λεπτό και κατόπιν στους σκιώδης εισηγητές για ένα τετράλεπτο για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Και αν απομείνει χρόνος θα μπορούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Θα δούμε ανάλογα με το χρόνο που θα μας μείνει διαθέσιμος πόσο χρόνο θα δώσουμε στους συναδέλφους και πόσο χρόνο θα έχουμε μέχρι τη μία παρατέταρτο. Κύριε Επίτροπε, εσείς πρώτα έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ähm, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ατουή, αγαπητοί εισηγητέ, κύριε και κύριοι βουλευτέ. Κυρίε και κύριοι ευχαριστώ για την πρόσκληση και Μπορώ να σας ε, παρουσιάσω τώρα τον προϋπολογισμό, την πρόταση προϋπολογισμού 2019, την οποία ενέκρινε μόλις ε, πριν από λίγα λεπτά το Σώμα των Επιτρόπων. Πρώτα απ' όλα σε εσάς, δηλαδή τον δημοσιονομικό μας έτερ. Και να σας παραπέμψω και στις 11 διαφάνειες τις οποίες μπορείτε να βλέπετε παράλληλα με την ομιλία μου. Η πρόταση αυτή προέκυψε κατόπιν σοβαρής ανάλυσης από την Κομισιόν και έτσι εφαρμόζουμε και μεταφράζουμε σε θέσεις του προπολογισμού τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Το σχέδιο αυτό του προϋπολογισμού βασίζεται στο υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και παρά την ε, προβλεπόμενη αποχώρηση των Βρετανών φίλων με βάση την μεταβατική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την σιγουριά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει στον προπολογισμό με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσει. Πρόκειται δηλαδή για έναν κανονικό εντό αγωγικών προπολογισμό των 28. Ε, πράγματι, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για τον τελευταίο προπολογισμό που θα εγκρίνει αυτό το Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι ο τελευταίο προπολογισμό που θα υποβάλει αυτή η Κομισιόν, γιατί σε ένα έτο ακριβώ. Λίγε ημέρες πριν από τι εκλογέ, θα πρέπει να παρουσιάσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο του 2020. Και Ελπίζουμε κατόπιν με το επόμενο κοινοβούλιο να εγκριθεί γύρω στον Οκτώβριο του 2019. Σας προτείνουμε για την ε, ανάληψη δαπανών να δεχτείτε ένα ποσό των 165 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα ποσό το οποίο έχει αυξηθεί κατά 3,1%. Ε, προτείνουμε ένα περιθώριο 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και για πιθανές εξελίξεις που αυτήν την στιγμή είναι απρόβλεπτες. Για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε γεωπολιτικές εντάσεις ε, και πιθανές στρατηγικές κινήσεις τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ τα μέσα ευελιξίας. Για το επόμενο έτος προτείνονται εδώ πέρα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε έχουμε μια αύξηση 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πάνω από το πλαφόν. Για τις πληρωμές προτείνουμε ένα ποσό 148,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι μια αύξηση 2,7% σε σχέση με το τρέχον έτος και μας αφήνει ένα αρκετά μεγάλο περιθώριο από 10,3 δισεκατομμυρία ευρώ μέχρι το ανώτατο όριο των δαπανών. Και βεβαίως αυτό οφείλεται στα γεγονότα των τελευταίων ετών γιατί βλέπουμε πως απαιτήθηκε μεγάλη ευελιξία για τα μέσα των πληρωμών. Κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου την Άνοιξη ήταν σαφές ότι Συμβούλιο Κοινοβούλιο και Κομισιόν έχουν μια συμφωνία όσον αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Στην πρότασή μας αναφέρουμε δύο τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη με δηλαδή για πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν επί σειρά ετών και ήδη μας απασχολούν εδώ και κάποια χρόνια. Πρώτον, η ενίσχυση της οικονομίας μας και της αγοράς εργασίας και η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνουμε μεγάλες αυξήσεις για κάποια προγράμματα κλειδιά που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, την δημιουργία θέσεων εργασίας και θα έχουν στο επικεντρό τη νέα γενιά. Και δεύτερο σημαντικό κομμάτι, μετανάστευση και ασφάλεια. Θα πρέπει, εφαρμόζοντας την αρχή της αλληλεγγύης, να δούμε το θέμα της μετανάστευσης και τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων με ιδιαίτερη έμφαση στα εξωτερικά σύνορα και εκτός της Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές και τις αιτίες τους, να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την σταθερότητα. Και ο προϋπολογισμός αυτός βεβαίω πάντα συμφωνεί με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης και πάντα μιλάμε για μέτρα που έχουν ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Έρχομαι στον τίτλο 1α, στην τέταρτη διαφάνεια. Το 1α περιλαμβάνει τις σημαντικότερες επενδύσεις για την ενίσχυση της οικονομίας μας και των θέσεων εργασίας. Προβλέπει 22,9 δισεκατομμύρια, μία αύξηση κατά 3,9% σε σχέση με τον προηγούμενο έτος. Μιλάμε για σημαντικές αυξήσεις για πολλά σημαντικά προγράμματα. Σε συμφωνία και με τον δικό σας μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Ορίζοντας 2020, τον οποίο, στον οποίο θέλουμε να δώσουμε 10,4 δις, αύξηση κατά 1 δις, πάνω από 8% δηλαδή. Το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, αύξηση κατά 1 δις στα 3,8 αύξηση 36% στον τομέα της καινοτομίας για να αυξηθεί αυτή η δυνατότητα στην Ευρώπη επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Υπάρχει εκεί πέρα το κοινό εγχείρημα για ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές. Και έχουμε ένα ποσό 194 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο έτος. Βεβαίως αυτά τα ποσά είναι μια αρχή, γιατί όταν μιλάμε για υπερυπολογιστές μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία απαιτούνται. Πρόκειται λοιπόν για ποσά τα οποία θα σωρευτούν στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η ψηφιακή Ευρώπη προτείνουμε ένα ποσό 9 δισεκατομμυρίων εκεί πέρα. Και εκεί λοιπόν θα δούμε τι μπορεί να γίνει για να δοθεί έμφαση ακριβώς στους υπερυπολογιστές. Το ίδιο επίσης ε, ενισχύεται και το θέμα της άμυνας, το οποίο έρχεται στο προσκήνιο. Και χαίρομαι ιδιαίτερω για την ε, συμφωνία χτες το βράδυ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου επί του θέματος. Έχουμε μια νέα πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας. Μιλάμε για 245 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προτείνουμε και έχουμε πάλι 25 εκατομμύρια για την προετοιμασία αυτών των μέσων. Και βεβαίως εδώ πέρα μας βοηθάει και ο χτεσινός συμβιβασμός. Είναι όλα επίσης παραμένει στο επίκεντρο. Τα μέσα για τον έρασμο συν αυξάνονται πάνω από 10%, 2,6 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι ένα βήμα προς μια κατεύθυνση που θα ενισχυθεί στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο ανέπτυξε πέρσι ως πρόταση η Κομισιόν και το οποίο ακόμα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, προβλέπουμε αυξημένα κονδύλια 100 εκατομμυρίων έτσι δημιουργείται μια βάση για να μπορέσουν χιλιάδες νέοι να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό έργο. Ελπίζω λοιπόν να εγκριθεί προσεχώς η νομική βάση από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί νομικά και δημοσιονομικά. Όσον αφορά την νεολαία, έχουμε το κομμάτι της πρωτοβουλίας απασχόλησης το οποίο είναι 233 εκατομμύρια ευρώ το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε και θα χρηματοδοτεί από τον τίτλο 1β. Αυτό πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα της οικονομικής ανάπτυξης γιατί έχουμε υψηλή ανεργία των νέων αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε σύγκριση με το 2013 η ανεργία των νέων από 24% τότε έχει πέσει σήμερα στο 15,6%. Και συμπληρώνουμε δυστυχώς στην εκτέλεση των προγραμμάτων, στην χρήση των κονδυλίων ακριβώς εκεί όπου είναι μεγαλύτερη η ανάγκη, στα κράτη-μέλη και περιφέρειες έχουμε χαμηλή πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή. Κάποια κράτη-μέλη έχουν τα χρησιμοποιούν τα κονδύλια που έχουν στην διάθεσή τους και δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό το οποίο υπάρχει, δυστυχώς. Ως Κομισιόν πριν από μερικές εβδομάδες ε, υποβάλα μια πρόταση για μια ευρωπαϊκή αρχή ε, εποπτείας της εργασίας που θα ασχολείται με την εσωτερική αγορά. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση εδώ πέρα για 11 εκατομμύρια ευρώ. Έρχομαι τώρα στην επόμενη σελίδα, τίτλος 1β. Ο τίτλος αυτός περιλαμβάνει και επενδύσεις για την πρόθεση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Και εδώ στο κύριο Βάρος εδώ πέρα πέφτει στα κράτη-μέλη. Η νέα γενιά προγραμμάτων και εφαρμογή τους, όπως ξέρετε, ξεκίνησε αργότερα από ό,τι περιμέναμε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πέρσι, τέλος ε, του 17, αυξήθηκε ο ρυθμός των πληρωμών. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά είναι μια θετική εξέλιξη. Και αυτό μας ε, κάνει να ελπίζουμε ότι δεν θα επαναλάβουμε τις άσχημες επιδόσεις της προηγούμενης φοράς. Στα τέλη του 17, όπως σας είπα, φτάσαμε σε πλήρη ταχύτητα και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και να ενισχυθεί φέτος. Εδώ, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Αυτό είναι άλλωστε και προς το συμφέρον των κρατών μελών. Ελπίζω λοιπόν ότι ο φιλόδοξος προϋπολογισμός πληρωμών δεν θα περικοπεί φέτος. Βλέπετε εδώ πέρα ξεκάθαρα στην διαφάνεια την εξέλιξη των προγραμμάτων από το 2007-2014 και βλέπετε την σταθερή άνοδο των πληρωμών. Ε, βλέπετε ότι εξαντλούνται τα προγράμματα του 2007-2013 και αυξάνονται τα προγράμματα του 2014-2020. Η πρότασή μας λοιπόν για τις πληρωμές περιλαμβάνει 47,1 δισεκατομμύρια ευρώ, μια ελάφρια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και αυτή η αύξηση μπορεί να φαίνεται μικρή, είναι αποτέλεσμα όμως της σαφούς μείωσης της ζήτηση για το προηγούμενο πρόγραμμα που βλέπετε ότι τίνει προς το 0 και της αύξησης για το τρέχον πρόγραμμα. Τα παλαιά προγράμματα θα εκπνεύσουν το 2019. Πρόκειται λοιπόν για το τελευταίο έτος στο οποίο υπάρχουν πληρωμές για την περίοδο 2007-2013 και έχουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά. Αν κοιτάξετε τα νέα προγράμματα, θα σημειώσετε αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2018, για το 2018, σε σχέση με το 2018, με βάση τα όσα προβλέπουμε ότι θα χρειαστεί να δαπανηθούν και να ε, μπουν στο αποθεματικό. Ωστόσο, τμήμα 2, γεωργικά προγράμματα σε σχέση με την συνοχή εδώ, μάλλον αντίθετα από τη συνοχή, είναι σχετικά σταθερά τα ποσά. Έχουμε 60 συνολικά δισεκατομμύρια, 1,2% αύξηση. Για το περιβάλλον όμως και τα μέτρα τα σχετικά με το κλίμα στο πλαίσιο του LIFE θα δείτε σημαντικότερη αύξηση, μεγαλύτερη του 8%. Μια εξέλιξη θετική που δείχνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος, από την κλιματική αλλαγή θα λάβει και, και την επόμενη χρονιά μεγάλη σημασία. Και βέβαια με βάση και τα όσα εσείς προτείνατε και ζητήσατε στην αρχή αυτής της περίοδου. Επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε το στόχο του 20% στις επενδύσεις για την προστασία από την κλιματική αλλαγή. Είχαμε μια σημαντική ακρόαση στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα στο θέμα αυτό. Αυτό το 8 και πλέον της 100 το πλησιάζουμε όλο και περισσότερο. Και επισημαίνω ότι για το επόμενο πούδου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο στο θέμα της κλιματικής αλλαγής προτείνει ένα 25% οριζόντιο ε, για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Εγκάρσια δηλαδή ώστε να καλύπτεται σε όλα τα προγράμματα. Στο, στην επόμενη διαφάνεια, στη διαφάνεια παριθμών 7, θα δείτε ότι οι προκλήσεις για το άσυλο και τη μετανάστευση μας υποχρεώνουν να λάβουμε δράση και να ενισχύσουμε την προστασία των συνόρων μας. Και έτσι λοιπόν στο τμήμα 3, ασφάλεια, ηθαγένεια, Βλέπετε τα σχετικά μέσα στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια βελτίωση και έχουμε λάβει υπόψη βέβαια τις προτάσεις του Κοινοβουλίου 360 εκατομμύρια ευρώ για την επαλήθευση του κανονισμού του Δουβλίνου, 175 εκατομμύρια για τη συνέχιση της βοήθειας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του ασύλου και το Ταμείο, και το Ταμείο Μετανάστευσης και ενσωμάτωση. Και τρίτον, έχουμε τα 117 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία, ε, πολιτική προστασία, προστασία από φυσικές καταστροφές. Αυτά είναι, αυτές είναι οι προτάσεις μας ε, που είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Επίσης, στο, σημείο, στο τμήμα 3, το συνολικό ποσό, και θέλω να το επισημάνω αυτό, ξεπερνάει το πλαφόν κατά 927,5 εκατομμύρια. Αυτή τη την ε, υπέρβαση μπορούμε να τη χρηματοδοτήσουμε μόνο χάρη στο μέσον ευελιξίας. στην κεφάλαιο υπαριθμών 8 τα μέτρα εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τμήμα 4 δηλαδή. Εδώ έχουμε σημαντικά νέα μέσα και δαπάνες σχετικά με την μετανάστευση, 13,1% αύξηση των ποσών για να φτάσουμε στο 11, στα 11,4 δισεκατομμύρια. πολύ περισσότερα από ότι το 2018 σε επενδύσεις για το θέμα αυτό και εδώ έχουμε το ε, καταπίστευμα για τους πρόσφυγες ε, σε ιδιαίτερη θέση. Ξέρετε ότι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα, ε, η πρώτη φάση, με πληρωμές που ξεπερνούν τα δύο δις και πλησιάζουν τα τρία. Και εδώ κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επισημάνω ότι συμφωνεί με το Συμβούλιο δεν υπάρχει. Αλλά Θέλω να καταλάβετε και εσείς ότι προσπαθώ σε κάθε συνεδρία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να είμαι πάντα παρόν σε αυτά τα θέματα. Το κύριο Συμβούλιο όμως συνεδριάζει κάθε ε, εβδομάδα με το Κορεπέρ, πιο συχνά από ότι το Κοινοβούλιο. Και πάω, αφού με προσκαλούν πάω. Και κάθε μέρα να με προσκαλούσαν πάλι θα πήγαινα. Και, σε, εσείς το ίδιο βεβαίως, νύχτα και μέρη με στη διάθεσή σας. Έχω αρκετή ε, αντοχή, αντοχές να ε, δουλεύω συνέχεια και τον Αύγουστο εδώ φάμε. Αν λοιπόν συνεδριάζει το Κοινοβούλιο και με προσκαλεί ή τους γενικούς μου διευθυντές ή τον συνάδελφο Χάν ή εμένα, θα πάω και εκεί γίνεται συζήτηση και Εάν με καλέσετε εσείς και μάλιστα μια μέρα πριν από το Κορεπέρ, πάλι θα είμαι εδώ και θα είμαι πιο συχνά από το Συμβούλιο. Το θέμα λοιπόν δεν είναι εάν είμαι διαθέσιμος να έρθω με συνεδριάσεις, αλλά πότε γίνονται συνεδριάσεις. Αυτό εξαρτάται μόνο από το δικό σας τον σχεδιασμό. Όπως είπαμε στη διάθεσή σας και στο Κορεπέρ. Έχουμε κάνει μία πρόταση, όπως έχουμε κάνει και σε εσά για τη δεύτερη αυτή φάση, για τα 3 δισεκατομμύρια. Και είναι κάτι επίγουσα η ανάγκη να αποδεσμευτούν τα ποσά αυτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χρειάζονται 8.000 δάσκαλοι και δασκάλες. Χρειάζεται αυτή η συμφωνία να έχει κλείσει πριν από τι θερινέ διακοπέ για να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Έχουμε δύο εκατομμύρια πρόσφυγε και των οποίων προσπαθούμε να δώσουμε στους οποίους προσπαθούμε να δώσουμε ε, για αυτούς και για τα παιδιά τους συνθήκες ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και αυτό για τα παιδιά σημαίνει σχολείο. Έχουμε συμφωνήσει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει το δρόμο τη προσφυγιά για να έρθουν στην Ευρώπη να του κρατήσουμε εκεί που είναι και να του εξασφαλίσουμε συνθήκε αξιοπρεπή. Χρειάζονται λοιπόν μετά το φαγητό, το νερό, τη στέγη, τη θέρμανση και την εκπαίδευση για τα παιδιά του. Εκεί που βρίσκονται πρέπει να διατεθούν αυτέ οι υπηρεσίε Και χρειάζονται, του ζητούν του δασκάλου το ταχύτερο δυνατό και χτε να του είχαν, θα του θέλανε και σήμερα και αύριο είναι σχεδόν αργά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για να συνάψουμε τη σχετική σύμβαση για κάθε σχολείο που χρειάζεται. Ένα δι σημαίνει αυτό από, τον Ευρωπαϊκό το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο και δύο επιπλέον δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα. Αυτό δυστυχώ, ξαφνικά το απέρριψε το Συμβούλιο πριν απο μηνε μήνες 7-8 κράτη-μέλη που τα γνωρίζετε κράτη-μέλη τα οποία εξαντλούνται σε εκλογικέ περιφέρειες, τα οποία συγγνώμη είναι στι εκλογικές σας περιφέρειες και τα γνωρίζετε καλά, αποφάσισαν ότι πρέπει όλα να βγουν από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Πράγμα το οποίο εμεί αδυνατούμε να εκτελέσουμε και να δεχθούμε. Ούτε κι εσείς βέβαια το δέχεστε. Αλλά απόφαση του Συμβουλίου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση του Συμβουλίου. Λοιπόν, το μόνο που έχουμε είναι η καταγραφή μιας ενδιάμεσης κατάστασης μέχρι που έχουν προχωρήσει δηλαδή οι συνομιλίες που ε, μόνο, το μόνο που δίνουν ότι το Συμβούλιο μπορεί, θα μπορούσε να δεχθεί ένα δισεκατομμύριο μόνο φρέσκο χρήμα. Και άρα ζητάει τα δύο δις να προέρθουν από αναδιανομή ποσών ε, του πουδουπού, του υφισταμένου πουδουπού. Αλλά επιπλέον. Το Συμβούλιο θέλει να παρέμβει ακόμα πιο πολύ στον τρόπο λειτουργία και να επιβάλλει από πού θα έρθουν αυτές οι αναδιανομέ για τα 700 τουλάχιστον εκατομμύρια. Αυτό θα μπορούσε να ληφθεί με απόφαση του Συμβουλίου, αλλά η Ιταλία δεν συμφωνεί. Βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση η Ιταλία, το γνωρίζετε φαντάζομαι και από τα όσα διαβάζετε στις εφημερίδες. Έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, αναμένεται να συναυθεί ένας νέος κυβερνητικός συναψηφισμός ακόμα και μέσα στη βδομάδα. Αυτό περιμένουμε. Αλλά εντολή από το Συμβούλιο, όσο δεν έχει δώσει την έγκριση της Ιταλία δεν μπορεί να υπάρξει. Μια ενδιάμεση πρόταση, ένα σχέδιο πρόταση που ενδεχομένω θα μπορούσε να δεχθεί το Συμβούλιο υφίσταται αυτή τη στιγμή και βεβαίω μετά μπορεί να περάσει και στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω μόνο να μην χρειαστεί να περιμένουν αυτοί οι γονεί και αυτά τα παιδιά ακόμα περισσότερε εβδομάδε. γιατί είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, είναι σημαντικό το θέμα, Βεβαίω με κάθε σεβασμό στη δυνατότητα σα να μελετήσετε και να συζητήσετε τα θέματα, αλλά πρέπει το αργότερο τον Ιούνιο να έχουμε απόφαση για αυτούς τους γονείς και αυτά τα παιδιά για να έχουν μια προοπτική για τον επόμενο χρόνο για τα σχολεία τους που είναι προτεραιότητα. Εμείς θα προτείνουμε 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2019 Και μπορώ να σας πω με ικανοποίηση ότι για το 2019 έχουμε διατηρήσει το 1,5 δις Και έτσι με τα μέτρα αυτά, τα δικά μας μέτρα, θα είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές να τις εκτελέσει πλήρως με βάση και τις ανάγκες όπως αυτές εντοπίζονται. το μέσον είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο γιατί ε, δίνει ε, χωρίς καμία παρέμβαση απευθείας ούτε της Άγκυρας ούτε κανένας άλλου Τούρκου Προέδρου Φερρυπίν ε, τα χρήματα στον όποιον τα έχει ανάγκη. Εδώ λοιπόν προτείνουμε 560 εκατομμύρια ευρώ για την δέσμευση όπως αυτή προέκυψε από τη Σύνοδο Κορυφής για την Συρία, και ακόμα ένα εκατομμύριο ευρώ για τη χρηματοδότηση μέσων και μέτρων για την οδό της Κεντρικής Μεσογείου αλλά και αντίστοιχα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και πάω στη διαφάνεια παριθμών 9. Η επισκόπηση των προγραμμάτων όπως σας προτείνονται στο σχέδιο. Έχουμε 60 προγράμματα με βελτίωση έτσι ώστε να προάγεται περισσότερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, αλλά και να υπάρχει και μια αξιολόγηση μέσω πρόθεσμη, με αντίστοιχη ενημέρωση και δική σας, να είναι δηλαδή πολύ πιο ε, ευανάγνωστα, όπως τα χρειάζεστε εσείς τα προγράμματα, ε, και σε ένα ενδιάμεσο στάδιο. Για να το εξασφαλίσουμε λοιπόν αυτό, Έχουμε καταρχάς ετοιμάσει σύντομες επισκοπήσεις ή περιλήψεις των προγραμμάτων. Και στη διαφάνεια 10 για τις διοικητικές ε, δαπάνες. Θέλω καταρχάς και ξεκινώντας να πω ότι με ικανοποίηση βλέπω ότι ε, μπορέσαμε μέσα στο ισχύον πολιτές οικονομικό πλαίσιο να περιορίσουμε σε επίπεδο όλων των ε, θεσμικών οργάνων κατά 5% το προσωπικό και αυτό είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα αξιοπιστίας ε, για το προσεχές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι πάρα πολύ, είμαι πολύ ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δική του τη συμβολή. Ε, στις δαπάνες που δεν έχουν να κάνουν με προσωπικό, δηλαδή συντάξεις και μισθούς, έχουμε οδηγήσει, οδηγηθεί σε μια ονομαστική σταθεροποίηση, πάγωμα δηλαδή των τιμών, αύξηση, και εδώ αυτό αφορά, το πάγωμα αφορά πούμε, τις για τα κτίρια, ε, αύξηση έχουμε μόνο σε θέματα που έχουν να κάνουν με μισθούς λόγω της αναπροσαρμογής, μόνο όμως σε επίπεδο 2,5% για τις συντάξεις η αύξηση έρχεται στο 6,2% και εδώ κυρίες και κύριοι θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε πολύ σύντομα το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη σημαντική αύξηση των, ε, των δαπανών για τις συντάξεις στα επόμενα χρόνια. Γιατί η αύξηση 6,2% δεν είναι το τελευταίο ποσό που θα δείτε σε αύξηση. Θα φτάσουμε και στο 8% και στο 10%. Αυτό προβλέπω και βλέπω ότι όταν έρθει η ώρα να αγγίξουμε το 12 και το 14% τότε θα θέσουν ορισμένα κράτη-μέλη το ζήτημα του εις ε, κάλυψης των αυξήσεων στις συντάξεις, του κόστου των συντάξεων, με την ε, περικοπή μισθών, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να δούμε. Είμαι λοιπόν πάντα σε άτυπες συνομιλίες ε, σε, ένα, σε επίπεδο στρογγυλής τραπέζης ενός συνταξιωτικού ταμείου το οποίο θα μπορέσει να καλύψει την αύξηση αυτή. Τώρα για να προχωρήσω στη σελίδα 11 και την επισκόπηση ο προπολογισμό του 2019 και σε αναλήψη υποχρεώσεων αλλά και σε πληρωμέ, όπω βλέπετε, σημειώνει πολύ ήπιε αυξήσει, περιορισμένε αυξήσει, απαραίτητε αυξήσει, με τι οποίε θέλουμε να ενισχύσουμε τι επενδύσει για την ανάπτυξη και την απασχόληση, που θα ενισχύσουν την εσωτερική δύναμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βοηθήσουν τα κράτη τα οποία υποδέχονται πρόσφυγε. Θα ενισχύσουμε την ευελιξία και τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να επισημάνω του δημοσιονομικού προγραμματισμού έχουμε αντιμετωπίσει δαπάνες, ανάγκες για δαπάνες, τελείως απρόβλεπτες λόγω των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και των φυσικών καταστροφών που αντιμετωπίσαμε. Στις 2 Μαΐου καταθέσαμε, μάλλον ετοιμάσαμε το σχέδιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα λύσουμε στις επόμενες εβδομάδες τους διάφορους τομείς. Μην ξεχνάμε όμως ότι και αυτός ο προϋπολογισμός του 19 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ να μας αφήσετε το περιθώριο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, όπως προβλέπετε, όπως προγραμματίζουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε έτοιμοι με τον προπολογισμό του 2019 και να τον εγκρίνουμε ε, όπως τακτικά προβλέπεται παρά την πίεση των ε, επερχόμενων ευρωεκλογών. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ακούσαμε τη, τις παρατηρήσεις και είμαστε έτοιμοι να προβλέψουμε νέες συνεδριάσεις. Πάντως, α, αν τα κανονίζετε όντω με το Συμβούλιο και όλα γίνονται στο Συμβούλιο, θα προτιμούσαμε το Συμβούλιο να έχουμε πιο συχνές επαφές για να μεταβιβάσουμε τις ανησυχίες μας. Ο χρόνο πιέζει. 7 λεπτά για τον κύριο Βιώτη. Ερωτήσει και απαντήσει. 4 λεπτά για τον Πολ Ρούμπιχ τα λοιπά τμήματα. Σκιώδη ηγητέ. 4 α, λεπτά καθένα. Έτσι φτάνουμε στα 37 λεπτά. Μετά ο κύριο Μούρεσαν για το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Έτσι θα έχουμε φτάσει στο 40 λεπτό. Αν όλοι τηρήσετε πιστά το χρόνο αγόρευσης θα τα καταφέρουμε. Θα είμαι πάντως αδιάλακτος, άτεγκτος. Κύριε Βιώτη, 7 λεπτά. 7 λεπτά που καλύπτουν τις δικές ερωτήσεις και τις απαντήσεις του Επιτρόπου. Οπότε αν θέλετε να λάβετε απαντήσεις, φροντίστε να ε, ολοκληρώσετε πριν το 7 λεπτό εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ξεκινώ ευχαριστώντας βέβαια τον Επίτροπο για την αυρόφροσύνη για το ότι ήρθε να μας ε, παρουσιάσει τον προϋπολογισμό χωρίς καθυστέρηση. Νομίζω ότι αυτό είναι και μια χειρονομία σεβασμού προς την Επιτροπή μας. Θέλω να το υπογραμμίσω και να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε. Και για να αυτό κι εγώ. Μην υποτιμάτε τη δική μας δυνατότητα να δουλεύουμε αδιάκοπα κύριε Επίτροπε. Είμαστε ικανοί να εισαγάγουμε στον προγραμματισμό μας και άτυπες και επίσημες συνεδριάσεις άπειρες. Σημειώνω λοιπόν περισσότερο παρά τίποτα άλλο τις παρατηρήσεις σας. Τα καταγράφω λοιπόν. Ασφαλώς θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να είμαστε έτοιμοι να διατυπώσουμε πιο λεπτομερή ζητήματα. Αλλά έχω τρία θέματα στα οποία θα ήθελα να διατυπώσω γενικές σκέψεις και να δω τις απαντήσεις σας. Καταρχάς το χρονικό ζήτημα, γιατί και εσείς το θίξατε και ο, Επίτροπος, και ο Πρόεδρος Αρτσουή και το μέσον για την Τουρκία. Πώς σκοπεύετε λοιπόν μέσα να βρείτε μέσα για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση αυτού του ε, μέσου του καταπιστεύοντος για την Τουρκία για το 19. Έχετε κάποιες ε, πιο λεπτομέρειες πληροφορίες να μας δώσετε και επίσης για να συμπληρώσω τα όσα είπε και ο Πρόεδρος γιατί παρά τις πιο τακτικές επαφές με το Συμβούλιο δεν κατατέθηκε ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού στην, ε, στον προϋπολογισμό του 2018 και για το θέμα της Τουρκίας. Κάτι ακόμη. με πολύ γενικέ σκέψει, όπω είπα, μετά θα κοιτάξουμε το σχέδιο του προπολογισμού στι λεπτομέρειε του. Ε, είπατε ότι κάνατε σεβαστέ τι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου, όπω τι είχαμε τον προηγούμενο Μάρτιο εγκρίνει με τα καταφυτηρίε γραμμέ. Και ιδιαίτερα ε, προτάει ένα προπολογισμό στρεφόμενο προ του νέου, τα μεγάλα προγράμματα που αφορούν του νέου, δηλαδή την Youth Initiative, πρωτοβουλία για του νέου και το Erasmus Plus. Μας προτείνεται ένα πρόγραμμα με κάποιες αυξήσεις, αλλά, και το λέω αυτό αμέσως, θα χρειαστεί περισσότερη δουλειά, κύριε Επίτροπε. Ο προπολογισμό και με τα περιθώρια που μα παρουσιάζεται μα επιτρέπει νομίζω να δουλέψουμε περισσότερο για να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη χρηματοδότηση για του νέου. Άλλωστε, εμεί στι κατευθυντήριε γραμμέ μιλούσαμε για ένα Erasmus Plus το οποίο και με βάση τις ιδέες που είχε προτείνει ο πρόεδρος Αρτουή θα διεύρυνε πολύ το φάσμα των δικαιούχων. Και, για, και το τρίτο θέμα κύριε Βίτροπε... μια πολιτική σκέψη, ελπίζω να μην έχω εξαντλήσει το χρόνο και να μπορέσετε να μου απαντήσετε. Σχέσεις με το Συμβούλιο. Όταν έρθει η ώρα για την συνδιαλλαγή, που είναι η πιο σκληρή και δύσκολη φάση, θα ε, επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Τώρα εσείς μας παρουσιάζετε έναν προϋπολογισμό που προβλέπει, ξέρω ότι θα, μπορούσατε να έχετε κάνει περισσότερα, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα πράγματα, αλλά έχετε σημειώσει κάποιες αυξήσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για, μες, για μας και στις αναλήψεις υποχρεώσεων και στις ε, πληρωμές και το θεωρώ θετικό αυτό. Ε, η ερώτησή μου λοιπόν έχει να κάνει με τις εντυπώσεις ε, που έχετε αποκομίσει σε σχέση με το Συμβούλιο. Τι περιμένετε δηλαδή ότι μπορεί να προκύψει από το Συμβούλιο σε σχέση με την ε, σύναψη συμφωνίας με βάση τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αλλά και αυτές που ορίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τις περιγράψατε σήμερα με το Συμβούλιο. είναι ο τελευταίο προπολογισμό. Ξέρω ότι πριν από τι προσεχεί ευρωεκλογέ θα μα καταθέσετε νέα πρόταση προπολογισμού, αλλά αυτό, ο προπολογισμό του 19 δηλαδή, είναι ο τελευταίο που θα εγκρίνει η τρέχουσα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Επομένω, θα ήθελα ε, να δω τι μπορώ να περιμένω για να αποκαταστήσουμε και την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι βέβαιο ότι μπορεί ο προπολογισμό να μα επιτρέψει να κάνουμε μια καλή δουλειά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε τι. Ε, μπορείτε να προβλέψετε για τη στάση του Συμβουλίου μας στους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε κύριε Βιώτη. Δύο λεπτά και δέκα δευτερόλεπτα έχετε κύριε Επίτροπε για την απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, Πρώτα απ' όλα για την ε, Τουρκία για το επόμενο έτος προτείνουμε ένα ποσό 1,45 δισεκατομμυρίων ως κομμάτι της επόμενης δόσης των τριών δις τα οποία όπως και στην ε, πρώτη δόση περιλαμβάνονται στο πρώτο εξεγόμεσο και στο πρόγραμμα ανθρωπιστικής Βοήθεια στον πρώτο πυλώνα με 850 δις και με 600 δις στον δεύτερο πυλώνα. Ε, εκατομμύρια με συγχωρείτε, αντιστοίχως 850 και 600. Και τα πιθανά δύο δις που θα μπορούσαμε συνολικά να ε, διαθέσουμε να καλυφθούν από 500 εκατομμύρια από το δημοσιονομικό έτος 2019 για να φτάσουμε στα 2 δις. Αναμένοντας πως τα κράτη-μέλη θα δώσουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο νέο χρήμα όπου τα κράτη-μέλη ήδη λένε πως δεν μπορεί να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 18 τον οποίων δεν θέλουν να αγγίξουν θα πρέπει να πάει στο 2019 και 20 στο Erasmus Plus για να το πω ξεκάθαρα Κοιτάξτε ε, όσο συμμετέχει ε, ένα τέσσερα ε, εκατό των φοιτητών κάθε έτος μπορεί να ανέβει πάρα πολύ. Μπορεί παραδείγματο χάρη να πάει από τα 30 στα 60 να διπλασιαστεί και να. Υπάρξει συνολικά μια αύξηση 10% ε, στα 2,6 δις συν 100 εκατομμύρια έξτρα. Στο Συμβούλιο νομίζω ότι θα είναι διαπραγματεύσει όπως και πέρσι, όχι ευκολότερε αλλά όχι και δυσκολότερες και μην ξεχνάμε ότι ε, βεβαίως ε, αυτά οφείλονται και στην ε, δική σας την χώρα. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο Πολ Ρούμπιχ για τα άλλα τμήματα του προπολογισμού. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερο στον Επίτροπο και την ομάδα του είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση κοιτώντα ε, το ότι προτείνεται 0,9% του ΑΕΠ νομίζω για το πολιτικό επίπεδο έχουμε ένα υποδειγματικό αποτέλεσμα 0,9% θα έλεγα ότι έχουμε ε, ένα πάρα πολύ οικονομικά συμφέρον θεσμικό όργανο. Βλέπουμε επίσης ότι εφαρμόστηκε η μείωση του προσωπικού κατά 5%. Θα ήθελα να δω συγκεκριμένα νούμερα όμως για το τι γίνεται και στα κράτη-μέλη. Γιατί βεβαίως αν είναι να λέμε ότι ε, αποτελεί υπόδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δούμε το τι γίνεται και στα κράτη-μέλη. Μιλήσατε για τις ε, συντάξεις και την αύξηση κατά 6,2% που αποτελεί ένα θέμα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θεωρώ πως η πρόταση ενός συνταξιωτικού ταμείου είναι η σωστή για να δούμε πώς θα ρυθμιστεί στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη ένα τέτοιο ταμείο το οποίο όμως ε, πλέον ε, δεν ε, χρηματοδοτείται, οπότε το ερώτημα είναι επειδή είμαι, είμαι και αρμόδιος για το τμήμα 2, γιατί έχουμε μία αύξηση κατά 18,5% στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασία Δεδομένων και 9% στον διαμεσολαβητή. Ενώ, παραδείγματο χάρη, το ελεγκτικό συνόδριο έχει δεκαδικά ψηφία, 0,5% είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις για τις εκτιμήσεις αυτή την φορά ήταν πολύ εκτεταμένες και θα με ενδιαφέρει να μάθω πώς έκανε αυτές τις προσαρμογές η Κομισιόν και πού έγιναν οι μεγαλύτερες οικονομίες. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό και γενικώ επίσης το λεγόμενο κόστος της μη Ευρώπης, ε, τι δηλαδή θα κόστιζε στα κράτη-μέλη αν αυτά τα πράγματα γινόταν σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεγητά, κύριε Ρούμπιχ. Αναφέρεστε σε αυτές τις τρεις υπηρεσίες. Προστασία προσωπικών δεδομένων, διαμεσολαβητή, ο πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό και 30 δεύτερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, αν συγκρίνετε αυτές τις τρεις υπηρεσίες, δηλαδή προστασία προσωπικών δεδομένων, ελεγκτικό συνέδριο και διαμεσολαβητή, η υπηρεσία έχει σημαντική αύξηση των ποσών με τον νέο κανονισμό και βελτίωση της απόδοσής της για το διαμεσολαβήτη, την διαμεσολαβήτρια με την οποία και μίλησα έχει τεράστια αύξηση υποθέσεων που φτάνουν στο γραφείο της. Και άρα χρειάζεται τη σχετική αύξηση προσωπικού. Και στις δύο όμως αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για μία ή δύο θέσεις προσωπικού. Όταν έχουμε να κάνουμε μια υπηρεσία που έχει 10-12 υπαλλήλους, πώς θα το συγκρίνεται αυτό με το ελεκτικό συνέδριο που ζηταει δύο, δύο-τρει-τέσσερι θέσει και άρα έχει πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό σας το λέω για να μην υπάρχει παρεξήγηση σε σχέση με, τον απόλυτο αριθμό θέσεων που επιπλέον δίνουμε. Το ελεκτικό συνέδριο έχει ένα σταθερό ρυθμό υποθέσεων να διαχειριστεί. Ενώ η υπηρεσία προσωπικών δεδομένων και η υπηρεσία του διαμεσολαβητή ζητάει, ζητάν μία αύξηση προσωπικού μικρή, ε, όπως είπα μία ε, δύο θέσεις, αλλά μόνο ε, εφάπαξ, όχι διαρκώς. Πέραμε στους και οδησηγητές για τέσσερα λεπτά, Μόνικα Χολμάιερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα περιοριστώ και εγώ επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καταρχάς τις ευχαριστίες για την πολύ συγκεκριμένη παρουσίαση του προϋπολογισμού στο 1α, 1β χαίρομαι που βλέπουμε την αύξηση. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε πολύ πιο προσεκτικά τα συγκεκριμένα ποσά γιατί στο τμήμα 1α ξέρουμε ότι υπάρχει ε, ανάγκη να βελτιώσουμε την ε, χρηματοδότηση γιατί έχουμε εξαιρετικές αιτήσει που χάνονται για δεκαδικούς πόντους διαφορά σε 98,5 ο ένας, σε 98 πόντους ο άλλος και δεν μπορούν δυστυχώς να γίνουν δεκτοί για ενίσχυση και εδώ μιλούμε για το κόσμο, μιλούμε για τα προγράμματα της τεχνολογίας και της καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου έχουμε ποσοστά αποδοχής από 3 μέχρι 7 το πολύ 100 πράγμα το οποίο βεβαίως που καταλαβαίνετε για τον Ετούντα είναι τεράστιο πρόβλημα και επικοινής φορείας. Και για τα εξωτερικά σύνορα χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω την αύξηση για τη Frontex, για την ασφάλεια των εξωτερικών σύνορων. Η προστασία των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως θα πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Αλλά καθώς είμαι και εισηγήτρια στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση Τρομοκρατίας. Πρέπει να πω ότι από τις επαφές που έχω και από τα Υπουργεία Εσωτερικών και το, οι σχετικέ υπηρεσίες διαπιστώνω ότι υπάρχει αντίστοιχο αίτημα και προς την Europol, η οποία όμως αναγκάζεται να τα απορρίψει, να τα απορρίψει τα αιτήματα αυτά γιατί δεν έχει αρκετό προσωπικό. Επομένω πρέπει να κοιτάξουμε γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη δουλειά που κάνει η Europol. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε και αυτό να το στηρίξουμε. Αναπτυξιακή βοήθεια επίσης. Προφανώς δεν μπορούμε πάλι να ζητούμε να μειωθούν κατά 50% τα κονδύλια που υποστηρίζουν τις χώρες αυτές από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες και μετά να ε, ξαφνιαζόμαστε γιατί ξαφνικά έχουμε μεγάλες δουλειές προσφύγων. Και εντάξει, έχουμε το καταπίστευμα το Ταμείο για την Τουρκία και πρέπει να δοθεί αυτή η υποστήριξη για τους δασκάλους και για τα 33.000 ε, παιδιά. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε. Για το τελευταίο, για τα 3 δισεκατομμύρια τα οποία εξαντλήθηκαν ήδη σε επίπεδο ανάληψης ε, δαπανών θα σας αποστείλουμε μια επιστολή με όλους τους αριθμούς τις επόμενες ημέρες των πρόεδρό σας. Οι πληρωμές εξακολουθούν να τρέχουν δεύτερον. Οι συνάδελφοι Νίμιτσα, Μογκερίνη και Χάν αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες ζωής ε, εκεί όπου κάνει έργα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, χειροτερεύουν, αλλά να περιορίζουμε τις αιτίε για τις οποίες φεύγει ο κόσμος. Και οπωσδήποτε στο επόμενο ΠΔΠ θα τα συζητήσουμε αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες. Το κόσμο είναι ένα πρόγραμμα για νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρές και μεσές. Πράγματι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και πολύ περισσότερα κονδύλια εδώ πέρα με τρόπο λογικό. Από την άλλη, βλέπετε ότι προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία όπου ε, μπορούμε. Βλέπετε ότι το λάθος εδώ πέρα ήταν ότι το 1,0 του ΑΕΠ σύνολο ήταν η βίβλος. Και υπάρχει η ΚΑΠ, η γεωργική πολιτική και η συνοχή, οπότε από κάπου έπρεπε να γίνουν περικοπές. Γι' αυτό ακριβώς οι δυνατότητες μας είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό ας μας γίνει μάθημα στην επόμενη φορά στο πρόγραμμα να μην περικόψουμε τόσο πολύ την πρόταση της ε, Κομισιόν για το κόσμο και την ψηφιακή Ευρώπη. Και θα το παλέψω αυτό τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλμερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Τιγκέρ. Ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση και τις πάντα εμπεριστατωμένες εξηγήσει που είναι βέβαια απαραίτητε για τα ποσά αυτά. Θα ξεκινήσω με ορισμένες παρατηρήσεις αλλά και ερωτήσεις. Αν και ξέρω ότι εμέσως μόνο είστε υπεύθυνος εδώ ε, για τα θέματα του προϋπολογισμού. Ε, γιατί είναι θέματα τα οποία πολιτικά αποφασίζονται και πρέπει να αποφασίζονται. Επί παράδειγμα, τη συμφωνία με την Τουρκία. Πριν από δύο περίπου χρόνια, σε μια κατάσταση ουσιαστικά έκτακτης ανάγκης, συνάψαμε μια συμφωνία με την ε, Τουρκία λέγοντα θα σας δώσουμε χρήματα. Και όλα αυτά μέσα σε συνθήκες ε, μεγάλης πίεσης. Και Βρισκόμαστε τώρα πάλι σε μια περίσταση όπου πρέπει πολύ γρήγορα πάλι να λάβουμε τέτοιου ειδου αποφάσεις και ρωτώ γιατί τέτοια πίεση χρονική. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια συνολική λύση για το μεταναστευτικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να γύρουμε και διαρωτώμε πόσο μπορούμε να πιέσουμε με μοχλό τον προϋπολογισμό τα κράτη-μέλη αλλά και το Κοινοβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί μια σαφής συγκεκριμένη βάση που θα δίνει μια μακροπρόθεσμη λύση στον τομέα αυτών του μεταναστευτικού. Επίσης, πολύ συχνά μιλούμε για την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας Τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το χρεολόγημα που έχω σήμερα ίσω να μην είμαι ο καταλληλότερο για να το συζητώ αυτό το θέμα αλλά στο θέμα αυτό τη ανθεκτικότητα, οπωσδήποτε πρέπει να συζητούμε τον ανταγωνισμό που βεβαίω ίσως δεν μπορεί να ε, αντιμετωπίσει κάθε δύναμη τη φύσης αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ε, πληθώρα επιχειρήσεων, εταιριών που μπορούν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, αλλά φαίνεται να θέλουμε να συγκρατήσουμε. Εμείς θέλουμε έναν ανταγωνισμό, ο οποίο θα επιτρέψει στον καθένα που έχει τη βούληση να αναπτύσσει τις δραστηριότητές του, να επιτρέπει ταυτόχρονα και την ανάπτυξη της οικονομίας και την θεκτικότητά Μπορείτε να πείτε κάτι σε αυτό, ο Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Βουλευτά. Την πρόταση για, το δεύτερο, για τη δεύτερη φάση, για το δεύτερο τμήμα, το, την κάναμε τον ε, Φεβρουάριο. Αλλά ξέρετε ότι η, τα γρανάζια αυτά προχωρούν και λειτουργούν πολύ αργά. Βεβαίως έχετε δίκιο, υπάρχει όλο αυτό το θέμα της ε, γειτονίας, της ευρωπαϊκής γειτονίας και το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στην περιοχή γύρω από την Ευρώπη σταθερότητα, ε, πώς μπορούμε ε, να ορίσουμε μια νόμιμη μορφή μετανάστευσης, μια ε, νομική βάση δηλαδή που θα εξασφαλίζει νόμιμη μετανάστευση. Όλα αυτά χρειάζονται προτεραιότητες σαφείς. Οι προτάσεις του κύριου Αβραμόπουλου, του συναδέλφου, για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προασύλου, της πολιτικής ασύλου, είναι ακόμα στο του Συμβουλίου, δεν τις έχει εγκρίνει. Επίσης, στο θέμα των μεταναστών. Χρειαζόμαστε 10.000 νέους υπαλλήλους για τις χώρες που κυρίως πλήττει μετανάστευση. Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, σε μερικέ περιπτώσει ακόμα και Πολωνία. Και ε, Ουκρανία για τη σταθεροποίηση. Χρειάζονται ε, έλεγχοι συνόρων και ενίσχυση των συστημάτων για την καταχώρηση των εισερχομένων. Στους να αναλαμβάνουν δραστηριότητα και είναι επιτυχή αυτή των κρατών μελών. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε στο προσεχέ πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια, παραδείγματι. Αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε. Το Ταμείο για την Αναπτυξιακή Βοήθεια μέσα στον, ε, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μια ιδέα η οποία νομίζω ταυτόχρονα ενισχύει και τη δική σα την αρμοδιότητα ε, οικονομία της αγοράς, ανταγωνισμός. Έχετε δίκιο βεβαίως, αλλά σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στον, ε, εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό από τις αμερικανικές και τις ιδιωτικές εταιρείε και εκεί πέρα είναι αδυσόπιτος ο ανταγωνισμός ε, και άρα πρέπει πάντα να εξασφαλίζουμε την θεώρηση του ναι μεν ελεύθερη οικονομία αγορά σε περιφερειακό επίπεδο αλλά ταυτόχρονα σε επίπεδο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και ανταγωνισμού στην βιοτεχνολογία, της, τα ηλεκτρονικά, τα, τη χαλιβουργία πολλές φορές είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις μας να αναπτύσσουν συμπράξεις και να ενισχύουν ε, μέσα από τη συνεργασία με και αμερικανικές εταιρείες μέσα, για, την, για όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά και της οικονομίας της. Ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε να ξεκινήσουμε μία φιλοφρόνηση. Χαιρετίζω την προσωπική σας προσήλωση στα δημοσιονομικά ζητήματα. Εκτιμούμε ιδιαίτερω τη συνεργασία με κάποιον τόσο ενθουσιώδη για τα θέματα αυτά και τόσο προσιλωμένο. Ε, τρία θέματα με προβληματίζουν. Δεν θα επισέλθω σε υπερβολικέ λεπτομέρειε. Πρώτη ερώτηση. Γενικώ, ε, οι προτάσει σα βαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μου. Και για μένα προσωπικά και για την ομάδα μου, η ακολουθούν τη σωστή άγουσα οι προτάσει. Παρόλο που για μερικά προγράμματα είναι κάπω ε, μικρό ο προπολογισμό, μιλήστε για το κόσμο, για άλλα. Πάντω, γενικώ οι προτάσει ε, θεωρούμε ότι είναι στη σωστή πορεία. Δεύτερον, τώρα είναι επαρκή τα μέσα που προβλέπετε. Η απάντηση είναι ε, αρνητική, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε και εσείς τίποτα, γιατί μας δεσμεύει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που μας βάζει τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθούμε. Τούτου λεχθέντος, έχω μία ερώτηση για τις πιστώσεις πληρωμών. Είδα ότι ε, είναι σοβαρή αύξηση στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θεωρείται όμως ότι η, η επιβάρυνση που θα έχουμε στο επόμενο πι δεν είναι υπερβολική, όπως συνέβη στην περίοδο 2014-2015 για το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα μετακυλθούν πολλά πληρωμές στο επόμενο. Επίσης, τα θέματα της μετανάστευσης. 175 εκατομμύρια ε, για την Ελλάδα. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση και με τους πρόσφυγες. Ε, αλλά δεν βλέπω τίποτα αντίστοιχο για την Ιταλία, τίποτα ειδικό για την Ιταλία. Ας μην ξεχνούμε την περίπτωση της Ιταλίας. Διάβασα στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που η πλειοψηφία του πληθυσμού θεωρεί ότι η χώρα δεν ε, έχει βγει κερδισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση η μοναδική χώρα που έχει τέτοια αρνητική γνώμη. Ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλοί που λένε ότι υποφελήθηκε η χώρα από την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην τελή πλειοψηφία θεωρεί ότι ε, δεν, ε, δεν βγήκε κερδισμένη η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν θέλουμε να έχουμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα με τον Brexit λόγω της δυσαρέσκειας των Ιταλών. Κύριε Πίτρο, έχετε το λόγο. Για την Ιταλία ειδικά πέρσι με τις δυνατότητες της ευελιξίας ε, υπήρχαν διάφορες έκτατες ε, χρηματοδοτήσεις όσον αφορά ζητήματα φυσικών καταστροφών, σεισμών, ε, αλλά και για την λεγόμενη δίωδο της Μεσογείου υπήρχε αξιόλογη στήριξη της Ιταλίας που θέλουμε να συνεχιστεί και φέτος. Αυτό το επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση της ε, χώρας. Παρ' όλα αυτά βεβαίως ε, το θέμα δεν είναι μόνο ζήτημα δικό μας, ε, είναι και ζήτημα της Ρώμης να εκταμιεύσει τα κονδύλια αντί να κατηγορούμε συνεχώς τις Βρυξέλλες. Πέρσι, στα ποσά είχαμε ε, ένα ποσό το οποίο ήταν στα 65,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν είχαν ε, ακόμα εκταμιστεί. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε ε, να κάνουμε τίποτα άλλο εμείς πέρα από τις εκκλήσεις και βεβαίως την άμεση εκταμίευση όταν ε, ζητείτε. Οπότε θα πρέπει να ληφθεί και μία απόφαση για το ύψος των δεσμεύσεων και των πληρωμών για το επόμενο ΠΔΠ για να ξεπεράσουμε αυτήν την φάση της ανασφάλειας. Και να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε απαντήσει τον Οκτώβριο για το θέμα αυτό των ε, ποσών αυτών που παραμένουν χωρίς να μιλούν. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Νεριάντα, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση και την ομιλία. Ε, νομίζω ότι ε, το πόσο καλός είναι ο προϋπολογισμός θα εξαρτηθεί από το πόσο εφαρμόζεται ε, και νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με την πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το κόσμο θέλουμε μεγαλύτερη ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βέβαια υπάρχουν άλλα, άλλες, άλλες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα, το Leisure Programming, είναι καλό, αλλά ε, είχαμε 13 μείωση σε 256 συνολικά εκατομμύρια. Ελάχιστα χρησιμοποίησαμε αυτή τη χρηματοδότηση. Πώς θα βελτιώσουμε λοιπόν την πρόσβαση των πολιτών σε τέτοια προγράμματα, γιατί είναι τελείω αποσυνδεδεμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτε. Θα πρέπει να προσθέσουμε τι διαδικασίε για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα διάφορα προγράμματα. Το ίδιο και το Erasmus Plus. Οι πιο εύποροι φοιτητέ μπορούν να υποφεληθούν από το Erasmus Plus. Οι οι λιγότερο εύποροι πρέπει να συνάψουν τραπεζικά δάνεια για να μπορέσουν να υποφεληθούν. Οπότε εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ε, το πώς θα εφαρμόσουμε καλύτερα τον προπολογισμό και θα βελτιώσουμε την πρόσβαση. Επίσης, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ανάπτυξης της ε, άμυνας στη βιομηχανία, πώς θα χρηματοδοτήσουμε αυτό το πρόγραμμα, μια και τα όρια του προπολογισμού είναι αρκετά στενά. Αυτά και ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βουλευτά. Συμφωνούμε ότι είναι πολλά τα προγράμματα ότι, όπου δεν, τα οποία δεν αξιοποιούνται γιατί είναι πολύ περίπλοκα. Και γι' αυτό προσπαθούμε με το Omnibus να εισαγάγουμε την απλοποίηση αυτών των κανόνων και στο προσεχές πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων το οποίο θα είναι ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρήσιμο γιατί αυτές είναι που φοβούνται την γραφειοκρατία περισσότερο και θα μπορούν έτσι να αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Βεβαίως, πολλές φορές έχει ε, επισημανθεί και από το Κοινοβούλιο το ζήτημα της καταστρατήγησης των κανόνων. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν απλοί κανόνες και για το Συμβούλιο και το Ελεκτικό Συνέδριο είναι πολύ σημαντικό ε, το ποσοστό του λάθους. Ε, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θέλουν ε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού την αδελφή Επιτροπή του ΣΥΠΗΝ. Ιδιαίτερα περίπλοκους κανόνες για να μην μπορεί να ξεφύγει τίποτε, για να έχουν κάθε λεπτομέρεια στη διάθεσή τους, αλλά βέβαια Πιστεύω τώρα θα έρθει η στην Κανά ελαφρύνει κάπως σε επίπεδο προπολογισμού για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Η απόφαση για την οποία με ενημέρωσε η κυρία Μπιερκόρσκα, η συναδελφός μου, μια απόφαση για την κατανομή κατά 50-50 στις αναδιανομές των ποσών, φρέσκο χρήμα και ε, αναδιανομές τώρα πάει σε ένα 60-40 60%, 60 φρέσκο χρήμα 40% αναδιανομές ή το αντίστροφο και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εξέλιξη η οποία από το 50-50 μας μεταφέρει σε ένα 60-40 και άρα το περιθώριο που έχουμε τα 60 εκατομμύρια περίπου θα πρέπει να το ε, ενσωματώσουμε στις νέες προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Τάραντ, Ίντρεκ Τάραντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με κάλυψαν ε, οι συνάδελφοι που είχαν την καλοσύνη να με προλάβουν, οπότε δεν χρειάζεται ούτε τι ερωτήσει να επαναλάβουμε, ούτε τι απαντήσει. Φυσικά δεν θα ήμουν μέρο των Πρασίνων αν δεν παραπονιόμουν ότι είναι ελάχιστα τα χρήματα για τις ε, πολιτικές ε, της συναφής με το κλίμα. Πάντως ευτυχώς ε, αυξήσετε κάποια σχετικά κονδύλια για το περιβάλλον και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Για το μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. γιατί να μην υποστηρίξουμε τις προτάσεις σας ό,τι αφορά το διορθωτικό προπολογισμό που βάλετε στο Συμβούλιο ε, από τη στιγμή που έγινε επίσημα αυτή η υποβολή. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές στα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η πιο συνετή, σοφή τακτική και έξυπνη τακτική εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να μην γίνει ο προπολογισμό ε, όμοιρο ή έρμεο του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και το αντίστροφο, γιατί είχαμε μια τέτοια εμπειρία στο παρελθόν. Πώ θα αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, ο τροποποιητικός προπολογισμό υπαριθμών 3 εγκρίθηκε σήμερα από εμάς. Αφορά πάλι την συμφωνία με την Τουρκία και ένα ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τις επόμενες ώρες ε, θα το λάβετε. Βεβαίως, Είναι προφανή η σχέση μεταξύ του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και του ετησίου προϋπολογισμού και βεβαίω το θέμα είναι ότι ο προϋπολογισμός του 14 και το δημοσιονομικό πλαίσιο 14 έως 20 διαπραγματεύθηκαν όλα μαζί το φθινόπωρο του 2013 και είχε παίξει το σημαντικό ρόλο ο κύριος ε, Σούλτς. Και βεβαίως ε, θα ε, χαιρόμουν να εγκριθεί εγκαίρως ο προπολογισμό του 19 εντός του 18. Και καλό θα ήταν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να μπορέσουμε να το εγκρίνουμε μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους. Ανεξαρτήτως των διαπραγματεύσεων για τον ετήσιο προπολογισμό. Γιατί τότε οι ερευνητέ, οι αγρότες, οι περιφέρειες, οι δήμοι θα γνωρίζουν το ύψος των ε, προσεχών προγραμμάτων. Και δεν θα υπάρχει έτσι η καθυστέρηση που υπήρχε το 14 και 15. Για μένα το ιδανικό θα ήταν Νοέμβριο του 18 να εγκριθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός και Μάρτιο του 19 το πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας και η τωρινή Κομισιόν τον Μάιο του επόμενου έτους να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τον ετήσιο προπολογισμό του 20 για να αποφασίσετε, δηλαδή το επόμενο Κοινοβούλιο, τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο και το Συμβούλιο και πιθανώς ή τρέχουσα Κομισιόν να αποφασίσει και αυτή με τη σειρά της ή πιθανώς η επόμενη. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Σίκφριτ Μούρεσαν, τον εισηγητή μας για τον προϋπολογισμό του 2018, για να σχολιάσει το τρίτο διορθωτικό προϋπολογισμό ε, για το 2018 και το μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Σύντομα όμως, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να σα δούμε και στην Επιτροπή Προπολογισμού, μια και είστε διαθέσιμο και πρόθυμο. Ο κύριο Μουρεσάν, σα ευχαριστώ και καλώ ήρθατε και πάλι. Χαιρόμαστε που σα ξαναβλέπουμε στην Επιτροπή μα. Καταρχήν, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού ε, που αφορά το μηχανισμό για του πρόσφυγε στην Τουρκία είναι από του σημαντικότερου που θα κληθούμε να ε, εγκρίνουμε ε, κατά το 2018. Γι' αυτό χρειαζόμαστε διαφάνεια. Ξέρω βέβαια ότι αυτό το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού σήμερα εγκρίθηκε στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε μόλις σήμερα. Επίσης, ε, θα δούμε πώς θα ε, χρηματοδοτηθεί το 2019. Μας το είπατε. Ποια είναι όμως η χρηματοδότηση του μηχανισμού αυτού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία για το 2018 ώστε ήδη να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε νοπό χρήμα, φρέσκο χρήμα, φρέσκους πόρους για το μηχανισμό αυτό και επίσης ευθυγραμμιζόμαστε με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα δισεκατομμύρια μόνο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και δύο δισεκατομμύρια από τα κράτη-μέλη. Η ερώτησή μου λοιπόν κύριε Επίτροπε είναι η εξή. Τι σας έκανε να αλλάξετε γνώμη σε σχέση με την αρχική σας πρόταση που τη βλέπαμε με πολύ καλύτερο μάτι. Βέβαια φαντάζομαι θα ήταν η άποψη του Συμβουλίου που σας έκανε να μεταπιστείτε. Ήταν μόνο η πολιτική πρόταση από το, πίεση από το Συμβούλιο που σας έκανε να αλλάξετε γνώμη ή κάτι άλλο για να αναθεωρήσετε την πρότασή σας ε, ε, στο διορθωτικό προϋπολογισμό. Από πέρυσι τον Οκτώβριο ε, είπαμε να συζητήσουμε το θέμα του μηχανισμού, ότι σίγουρα ε, και εμεί ήμασταν πρόθυμοι εδώ και καιρό να συνεργαστούμε. Την πίστη πρέπει να την κατευθύνετε προ το Συμβούλιο. Εμεί θα ήμασταν καθεν πρόθυμοι. Τα τελευταία δύο χρόνια πήγαμε στην Τουρκία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, στην Τινησία και όπω είπατε κι εσεί, για την παιδεία χρειάζεται κάποια προβλεψιμότητα. Το γνωρίζουμε, αλλά δεν φταίμε εμεί για την καθυστέρηση, το Συμβούλιο. Και είναι απαράδεκτο το Συμβούλιο να κολλησιεργεί και μετά να πιέζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελευταία στιγμή και άρον άρον να λαμβάνει τις αποφάσεις ενώ εμείς είμαστε ανέκαθεν πρόθυμοι για, τη... Ε, για τη συνεργασία. Και αυτά θέλουμε τώρα χρόνο στις πολιτικές ομάδες για να αποκρισταλώσουμε τις θέσεις μας. Ε, είπα ότι θέλουμε από το φθινόπωρο θα, να είμαστε έτοιμοι, αλλά αναρωτιόμαστε αν ήταν ειλικρινή το σχέδιο προπολογισμού για το 2018 δεδομένου ότι δεν ελειφθεί υπόψη ο μηχανισμός για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, δεν ήσασταν νομίζω νωρίτερα μια άλλη φορά που είχα έρθει, άρα κατά κάποιο τρόπο πρέπει να τα επαναλάβω. Όντως σήμερα Κάνουμε το διορθωτικό προπολογισμό. Τον συμφωνούμε σήμερα, τον τρίτο διορθωτικό για το 2018 και αυτό αναφέρεται στο ε, μέσον για την Τουρκία. 550 εκατομμύρια ευρώ για το 2018. ...500 εκατομμύρια φρέσκο χρήμα, συμπληρωματικά κονδύλια δηλαδή, ε, συμπληρωματική πόρη... ...και 50 από το earmarking, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια. Από τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας κάνουμε earmarking και εξασφαλίζουμε αυτά τα 50 εκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες μας συζητούν το ίδιο θέμα και το υποβάλλουν στο Συμβούλιο ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι είμαι αγγελιαφόρο λίγο πολύ. Θα μεταφέρω δηλαδή τι επικρίσει προ το Συμβούλιο. Θα το πράξω. Αλλά είμαι μέλο τη Επιτροπή και άρα σε περιορισμένο βαθμό μόνο υπεύθυνο σε σχέση με τα όσα καταγγέλλεται για το Συμβούλιο. Άρα βεβαίως θα μεταφέρω το, ε, την επίκριση ότι το Κοινοβούλιο και έχει δίκιο σε αυτό, καταγγέλει, κατακρίνει την ε, διεξαγωγή, τον ε, χρονισμό αυτών των προτάσεων και, ότι, και το γεγονό ότι εμείς, ενώ εμείς κάναμε προτάσεις τον Φεβρουάριο του 2018 έχουν μέχρι το Μάιο μείνει στο τραπέζι του Συμβουλίου οι προτάσεις αυτές έχουν μείνει σε αδιέξοδο και επειδή η Ιταλία δεν είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση δεν είναι σε θέση το Συμβούλιο να συνεχίσει τις συνομιλίες του. Και ξέρουμε ότι το Συμβούλιο αρνούνταν κατηγορηματικά να δώσει 2 δισεκατομμύρια επιπλέον. 7 κράτη-μέλη, μεγάλα κράτη-μέλη, Γερμανία, Γαλλία και λοιποί, μας κάλεσαν σε μια επιστολή ε, πέρσι την Άνοιξη να διαθέσουμε, να βρούμε μάλλον τα κονδύλια αυτά, τα τρία δις από αναδιανομές και φτάσαμε σιγά σιγά σε ένα συμβιβασμό που θα σήμαινε ότι θα μπορούσε το Συμβούλιο να εξασφαλίσει να δώσει ένα δισεκατομμύριο φρέσκο χρήμα. Ίσως θα μπορούσε να δώσει. Παραλαμβάνω, δεν είμαι εγώ αρμόδιος γι' αυτό. Για μας σημασία έχει το ταχύτερο δυνατό να ληφθεί απόφαση για τους ανθρώπους αυτούς, για τις μαθήτρες και τους μαθητές, για τα παιδιά που είναι στην Τουρκία. Καλώς. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της ακρόασης, κύριε Επίτροπε. Έπρεπε να φύγετε μία παρατέταρτο, είναι ήδη μία παραπέντε. Δυστυχώς οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν το λόγο. Θα ήθελα πάντως να σας πω ότι το σχέδιο προπολογισμού για το 2019 και το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμό 3 για το 2018 μόλις ε, σας απεστάλησαν ε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οπότε θα έχετε την ευκαιρία να εντρυφήσετε στις λεπτομέρειες αυτών των δύο σχεδίων και σίγουρα θέλουμε να ε, διεκπαιρώσουμε μέχρι το Μάρτιο του 2019 το, το, τις διαπραγματεύσεις ε, αλλά με 265 δις ε, υπόλοιπα προς εκαθάριση δεν θεωρείται ότι θα έχετε προβλήματα ταμιακά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξοφλήσετε τους προϋπολογισμούς του προηγούμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και αμέσως μετά να ξεκινήσετε το νέο ΠΔΠ. Θα μπορούσατε σε επόμενες εβδομάδες να μας κάνετε κάποιες προβλέψεις ε, για τις ε, ταμιακές ροές ώστε ε, να δούμε πώς θα καλύψουμε τα υπόλοιπα προσεκαθάριση επόμενη της προηγούμενης δημοσιονομικής περίοδου ώστε να ξεκινήσουμε την επόμενη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε πρώτα στην Επιτροπή Προπολογισμών πριν κάνετε τις δηλώσεις στον τύπο. Η συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου δυστυχώς ακυρώνεται, ξέρω πόσο σας απογοητεύει αυτό. Η επόμενη μας συνεδρία θα γίνει στις 18 Ιουνίου και αμέσως μετά 19 Ιουνίου, δηλαδή διήμερη συνεδρίαση 18 και 19 Ιουνίου. Αυτά και λίγα τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή.